rufe auf die stimmerklärungen zunächst zum entwurf des gesamthaushaltsplans der europäischen union für das haushaltsjahr. Τώρα περάσουμε ψήφου. Πρώτα απ' όλα σε ό,τι αφορά τον του 2010. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην εποχή που οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να κάνουν περικοπές στους προϋπολογισμούς τους και οι ε, πολίτες το ίδιο πόσο χαρακτηριστική είναι η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία αυξάνει τον προϋπολογισμό της. Τούτο θα έχει πολύ σημαντικές συνέπειες στις χώρες μέλη. Στη δική μου χώρα, παραδείγματο χάρη, η συνεισφορά μας θα αυξηθεί κατά 16% τους προσεχείς 12 μήνες. Για να το εξηγήσω, στο τελευταίο συνέδριο του κόμματό μας ε, δεχθήκαμε ότι θα κάνουμε περικοπές 7 εκατομμυρίων λιρών 7 δισεκατομμυρίων ε, λιρών ε, συνολικά. Από την άλλη βλέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχει ε, αυτή η γαλαντομία. Δηλαδή παίρνουμε από τα τσέπες των ανθρώπων και τα ξοδεύουμε για την διεύρυνση της γραφειοκρατίας. Αν ήταν τέτοια η συμπεριφορά μας στο παρελθόν θα είχαμε χάσει τον ε, ψυχρό πόλεμο. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται μόνο με την απασχόληση των υπαλλήλων της και γι' αυτό αυξάνει και διονγκώνεται ο προπολογισμό. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντότς έχει το λόγο, λέει ο Πρόεδρος. Frau Kollegin Dotz. Η κυρία Ντότς, θέλω να καταστήσω σαφές ότι υποστήριξα τις τροπολογίες 732 και 733 και είναι κρίμα που το σώμα δεν τις υποστήριξε. Χαιρετίζω οποιοδήποτε μέσο που ε, που βοηθάει στην μη κατάργηση των οικογενειακών προγραμμάτων που αφορούν την ε, ε, στήρωση κλπ. Επίσης, ε, ε, ε, επίσης θα πρέπει να χαιρετήσουμε όλες εκείνες τις προσπάθειες οι οποίες αφορούν την επιλεκτική γέννηση φύλου σε χώρες της Ασίας. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε υπέρ τέτοιων προγραμμάτων. Ευχαριστώ κυρία Ντότσο. Αυτέ ήταν οι επεξηγήσεις ε, ψήφου στο Γενικό Προπολογισμό 2010. Περνούμε στην έκθεση Surgeon. Η κυρία Ρότσαν έχει το λόγο. Θα ήθελα να πω και εγώ και πρέπει ότι λυπούμε που δεν μπορέσαμε να ψηφίσουμε υπέρ της αναπτυξιακής βοήθειας και ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε χρήματα ε, υπέρ του οικογενειακού προγραμματισμού και κατά των αμβλώσεων. Ξέρουμε ότι σε άλλες υπήρους, κυρίως στην Αφρική, είναι υποχρεωμένες οι γυναίκες να υποστούν έκτρωση εάν κυοφορούν ε, κορίτσια. Πιστεύω ότι θα πρέπει να στείλουμε χρήματα σε όσους υποστηρίζουν την κατάρριξη τέτοιου είδους ε, διακρίσεων. Και θα πρέπει τέτοιου είδου δικλείς ασφαλή να τι υπερψηφίζουμε όταν ψηφίζουμε τον προπολογισμό. Ευχαριστώ, κυρία Ρόιτεβα. Ο κύριο Μπόλτσο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εάν δείτε τις τροπολογίες, σε πολλές από αυτές θα δείτε ότι υπήρχαν ε, κάποια κομμάτια στο κείμενο που άλλαξαν εντελώς εξαιτίας της διατύπωσης το όλο κείμενο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την απόρριψη μιας σχετικής τροπολογίας απέδειξε ότι δεν έμαθε από τα παθήματα των τελευταίων ετών δεν κατάλαβε και δεν κατανόησε τι ακριβώς συνέβη από την ε, φιλελευθεροποίηση των αγορών. Νομίζω ότι δεν έμαθε ότι δεν πρέπει να συνεχίσουμε προς την ίδια κατεύθυνση. Βλέπουμε ότι εμείς συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τους ισχυρούς της νεοφιλελεύθερης αγοράς παρά το γεγονός ότι υπέστη μεγάλο πλήγμα το σύνολο της Ευρώπης, οι πολίτες της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκόλνης. Κύριε Πρόεδρε. Ενώ τα Ινστιτούτα διαφόρων προγραμμάτων που είναι προγράμματα που αφορούν ε, την ισχύουσα θέση κάποιων που ασχολούνται με την εκπαίδευση, με άλλα θέματα, δεν κάναμε τίποτα για να βοηθήσουμε τους γαλακτοκόμους. Είχαμε δύο τροπολογίες, την 812 και την 70. Η 812 με τη συμφωνία του Συμβουλίου προέβλεψε τη χορήγηση 300 εκατομμυρίων. Η 812 600 εκατομμύρια. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, είπαμε ότι την 70 θα ψηφίσουμε πρώτα. Και στο άρθρο 61, παράγραφο 2 του κανονισμού, λέει ότι αν δύο τροπολογίες που αυτοαποκλείονται αφορούν το ίδιο μέρος του κειμένου, αυτό που απομακρύνεται περισσότερο από το αρχικό κείμενο έχει την προτεραιότητα και πρέπει να ψηφιστεί κατά πρώτο λόγο. Ο εισηγητή ανέφερε έναν άτυπο κανονισμό, αλλά ο κανονισμό του Κοινοβουλίου έχει την προτεραιότητα και κάποιο χρησιμοποίησε αυτή τη διαδικασία και είναι σκανδαλώδες το ότι δεν ψηφίστηκε πρώτα απ' όλα έτσι όπως έπρεπε η τροπολογία η οποία αφορούσε τα 600 εκατομμύρια τους ε, γαλακτοκόμους. Ναι, έκθεση. Μάνκα. Συνάδελφος Πικοβίτσε. Aš balsavau už metų biudžetą, nes... Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας εξηγήσω ότι υπερψήφισα τον προπολογισμό 2010, δεδομένου ότι τα κονδύλια που έχουν προβλεφθεί θα διευκολύνουν την κατάσταση για τους πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται εξαιτίας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης σε δύσκολη θέση. Είναι για την παρούσα περίοδο πάρα πολύ σημαντικό αυτό, δεδομένου ότι λαμβάνουμε υπόψη και τις κοινωνικές ανάγκες των ατόμων. Υπερψήφισα επίσης τα κονδύλια που προβλέπταν για την δημιουργία θέσεων απασχόλησης και διατήρηση θέσεων απασχόλησης. Είναι επίσης εξίσου σημαντικό να έχουμε να προβλέψουμε κάτι για το γαλακτοκομικό τομέα. Θα μπορούσαμε να δώσουμε περισσότερα ε, κονδύλια στους γαλακτοκόμους, αλλά πάλι καλά που τους δώσαμε και αυτά που τους δώσαμε. Σας ευχαριστώ κυρία Πικαβιτσιούτε. Επόμενος ομιλητής, κύριος Φαντάλεν. Κύριε Πρόεδρε, εγώ καταψήφισα τον προϋπολογισμό, διότι όλες ε, τα κονδύλια αυξάνονται, εδώ όλες οι χώρες κάνουν κρατικούς προπολογισμούς όλο και πιο σφιχτούς. Δεν βλέπω γιατί κάνουν αυτό οι κρατικοί προπολογισμοί και εδώ όλο αυξάνουμε τα κονδύλια, αυξάνοντας και τους ε, απολαβές των ε, αξιωματούχων και όχι μόνον, ακόμη και άλλα επιδόματα κυρίως ε, για τα δαπάνε, για το τηλέφωνο, για την ε, γραφειακή υποστήριξη, ενώ κανένα δεν χρειάζεται να αιτιολογήσει γιατί χρειάζεται περισσότερα χρήματα. Τους δίνουμε λοιπόν μία επιταγή εν λευκό. Και για να σας πω, ε, αυτά τα οποία λέμε εμείς ε, στην Ολλανδία, δωράκι του Άγιου Βασίλη τους κάνουμε. Χωρί να ζητούμε λογαριασμό από κανέναν. Ελπίζω λοιπόν ότι οι συνάδελφοι θα σκεφτούν αυτό το δωράκι, το 242 ευρώ που πήρε ο καθένας, για να το χρησιμοποιήσουν με χρήσιμο τρόπο. Επεξηγήσεις ψήφου τώρα την... Ε, Πρώτα κανονισμού του Συμβουλίου 1234. Η κυρία Μολβάη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, υπερψήφισα τα μέτρα για να μπορέσει να βελτιωθεί η κατάσταση στον γαλακτοκομικό τομέα και θα ήθελα να πω το εξής. Αυτό που δίδουμε εδώ είναι ψίχουλα, είναι ελάχιστα ποσά. Ξέρουμε ότι δεν μπορεί να διορθωθεί η όλη κατάσταση. Δεν είναι καλύτερα να καταψηφίσουμε σε αυτό το ποσό. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι Τρία ερωτήματα έθεσα και δεν πήρα ακόμη καμία απάντηση. Τι προτίθεται να κάνει σε σχέση με την κρίση Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι πηδάμε από τη μία κράση, κρίση συγγνώμη, στην άλλη. Τι προτίθεστε να κάνετε, τι μαθήματα έμαθε από αυτήν την τραγική κατάσταση, αυτήν την καταστροφή των γαλακτοκόμων η Ευρωπαϊκή Ένωση που κατέστρεψε τη ζωή τόσων πολλών εκατομμυρίων ε, χιλιάδων συγγνώμη, νοικοκυριών. Πώς θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι τα κονδύλια που δώσαμε είναι κονδύλια από τα οποία θα υποφεληθούν πρώτα οι μικροί γαλακτοκόμοι και όχι τα μεγάλα εργοστάσια. Επίσης, τι θα κάνετε με τις ε, διακρίσεις που υπάρχουν ε, ε, κατά των νέων χωρών. Ευχαριστώ, ο κύριος Γιάρεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω τρεις παρατηρήσεις σε σχέση με τον γαλακτοκομικό τομέα. Χαίρομαι πρέπει να πω πρώτα απ' διότι αντέδρασε η Επιτροπή μετά τα διάφορα προβλήματα που είδαμε να αντιμετωπίζει ο γαλακτοκομικός τομέας. Επίσης, τα χρήματα δεν είναι το πάνι για να δοθεί μια κατάσταση. Πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο στο να σκεφτούμε πώς θα κάνουμε τη μεταρρύθμιση του τομέα αυτού. Θα ήθελα να υπάρχει διάλογος μεταξύ των επαγγελματιών του κλάδου αυτού και των ε, πολιτικών για να δούμε πώς μπορούμε να οργανώσουμε την ε, αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων μετά το 2015. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ρόιτοβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υποστηρίζω πλήρως την ε, ε, επέκταση της ισχύω του κανονισμού βάσει το άρθρο 176 για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε με ευέλικτο τρόπο στις ε, αλλαγές που πρέπει να υπάρξουν στο γαλακτοκομικό τομέα χωρίς να στρεβλώσουμε τις συνθήκες ανταγωνισμού. πρέπει να πω ότι όλοι οι κρατικοί προϋπολογισμοί δεν έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν τα μέτρα τα οποία προβλέπονται για τη στήριξη του κλάδου και πιστεύω ότι θα υπάρξουν στρεβλώσεις στην αγορά. Δεν θέλουμε να υπάρξει στρέβλωση της αγοράς και της ανταγωνιστικότητας. Εγώ προτιμώ η Ευρωπαϊκή Ένωση να διευθετήσει το θέμα των ποσοστώσεων και την ε, ίση πρόσβαση όλων στις αγορές. Γι' αυτό απήχα εγώ από αυτή την ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κίσκι. Κυρίες και κύριοι, μετά από στην Επιτροπή Γεωργίας και μετά από πολλές διαμαρτυρίες αγροτών στις χώρες μέλη, τελικά καταλήξαμε στην επιπρόσθετη υποστήριξη των γαλακτοπαραγωγών. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό, διότι οι άνθρωποι αυτοί έχασαν πολλά και οι περισσότεροι βρίσκονται στο χείλος της χρεοκοπίας. Επίσης η φήμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπονομεύεται. Για ποιο λόγο έδρασε τόσο καθυστερημένα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπήρχε αρκετή εποπτεία, επαρκής εποπτεία της αγοράς. Τούτο δεν είναι ε, πολύ θετικό ε, όσον αφορά τη λειτουργία της διοίκησής μας. Υπενθυμίζω ότι όταν καθυστερούμε οι ε, δράσεις που αναλαμβάνονται κοστίζουν πολύ περισσότερο. Πρέπει λοιπόν να σταθεροποιήσουμε τις αγορές και ιδιαιτέρως υπό τη σημερινή κατάσταση και να διασφαλίσουμε τη μακροπρόθεσμη ε, παραγωγή ιδιαίτερα έναντι αυτών των πολύ σκληρά εργαζομένων γεωργών. Ευχαριστώ κύριε Σεκέλσκι. Έχω άλλες δύο επεξηγήσεις ψήφου, λέει ο Πρόεδρος. Αλλά πρέπει να επισημάνω ότι σύμφωνα με το άρθρο 170 η επεξήγηση ψήφου δεν μπορεί να ζητηθεί από τη στιγμή που έχει αρχίσει η πρώτη επεξήγηση επί της εκθέσεως. Επειδή πρόκειται για νέα μέλη θα δεχθώ τώρα την παραβίαση του κανονισμού. Πρέπει όμως να τηρήσουμε την σειρά. Ο συνάδελφος Κένι έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Καταρχήν θέλω να πω ότι και εγώ χαίρομαι που εγκρίναμε τον επιπρόσθετη ενίσχυση για τους γαλακτοπαραγωγούς. Τούτο δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ακούει και αντιδρά προφανώς εντός των δυνατοτήτων που προσφέρει ο προϋπολογισμός. Θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε ακόμη περισσότερο τους ε, γαλακτοπαραγωγούς. Ελπίζω αυτό να γίνει στο μέλλον. Δεύτερον, στην αγγλική μετάφραση σήμερα έγιναν κάποια λάθη και ο κύριος Μπούζακ πολύ ευγενικά είπε ότι ίσως οφείλονταν στο ότι μιλούσε ο ίδιος πολύ αργά. Δεν θέλω να... Ε, δεν θέλω να επιτιμήσω κανέναν, ωστόσο πολλές φορές έγιναν λάθη στους αριθμούς, δηλαδή το 908 ελέγχθη ως 909, το 444 ως 445 κλπ. Παρακαλώ αυτό να ληφθεί υπόψη. Και βεβαίως δεν λειτουργούσε και ο, ο ηλεκτρονικός πίνακας. Και αυτό βεβαίως είναι ε, ηλεκτρονικό σφάλμα. Ε, ευχαριστώ κύριε Κέλλης. Ο κύριος Καλινόφσκι έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ ψήφισα υπέρ της τροπολογίας κανονισμού Ωστόσο έχω αμφιβολίες, διότι το νέο σύστημα υπολογισμού των προστήμων θα τεθεί σε ισχύ από 1η Απριλίου. Εν πάση περιπτώσει εγώ ψήφισα υπέρ διότι αυτή η αλλαγή δίνει τη δυνατότητα υποστήριξης των γαλαπαραγωγών με 280 εκατομμύρια ευρώ και μπορούμε να ελπίζουμε ότι η χειρότερη περίοδος έχει περάσει. Τίθεται το ερώτημα βέβαια θα, ποιο θα είναι το μέλλον της παραγωγής γάλακτος στην Ευρώπη και ιδιαίτερος πώς θα λειτουργήσει το σύστημα των ποσοστώσεων. Διότι αφενός έχουμε μια πρόταση για αύξηση των ποσοστώσεων ενώ από την άλλη υπάρχει πρόταση μείωσης της παραγωγής. Ευχαριστώ κύριε Καλινόφσκι και ερχόμαστε στο τέλος των επεξηγήσεων ψήφου επί του προϋπολογισμού του 2010 και τώρα, τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Χέν για τις εξωτερικές σχέσεις. Ο Ντεκάρτ έλεγε ότι ίσως χρησιμοποιούνται όλες οι αισθήσει μας από έναν κακό δαίμονα. Ε, μερικές φορές ακούγοντας ε, τους συνομιλητές εδώ, τους ομιλούντες, ε, αισθάνομαι ότι βρισκόμαστε σε μια εντελώς εξωκαρτισιανή κατάσταση. Ερχόμαστε τώρα στον πραγματικό κόσμο. Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ουσιαστικά υποστηρίζει τους τυράννους στο Πεκίνο ή απομονώνει την Ταϊβάν. Ε, υποστηρίζει τους κουβανούς ε, ηγέτες ή συνεργάζεται με τους ε, Αγιατολάχ ή αυτούς, την Χαμά στην Παλαιστίνη. Δηλαδή η, διάδοση της δημοκρατίας ε, με τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν καμία σχέση. Δεν λέω ότι δεν είναι δημοκρατική η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ασκούμε αυτά τα δικαιώματα εντός ε, της Ένωσης, ωστόσο στην εξωτερική πολιτική υποστηρίζουμε τέτοιες κυβερνήσεις και δεν επιδιώκουμε το ε, κράτος δημοκρατικού δικαίου το οποίο ε, υποστηρίζουμε. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος, ο κύριος Κάμαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν νομίζω ότι κανένας θα διαφωνήσει μαζί μου ότι χρειάζεται να υποστηρίζουμε και να προαγάγουμε τη δημοκρατία σε ολόκληρο τον κόσμο εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εντός αλλά θυμάμαι αν κοιτάξουμε ε, την ιστορία, θυμάμαι ότι όταν οι Ηνωμένε Πολιτείε προήγαγε τη δημοκρατία σε ολόκληρο τον κόσμο και τους λέγαμε «Μα τι κάνετε πίσω αυλή σας», δηλαδή τους ε, Αμερικανούς που στερούνταν τα ατομικά του δικαιώματα. Το ίδιο με τη Βρετανία. Στη Βρετανία η οποία επιδίωκε τη διάδοση της δημοκρατίας σε ολόκληρο τον κόσμο αλλά αρνούνταν την ψήφο στι γυναίκες. Και τώρα ε, το ίδιο κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο συνάδελφός μου ο κύριο Άννεν έδωσε πολλές λεπτομέρειες αυτή τη υποκρισία. Όταν μιλούμε για τη διάδοση της δημοκρατίας πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι τα δικά μας είναι σε απόλυτη τάξη και οι Γάλλοι και οι Ολλανδοί γνωρίζουν πολύ καλά το τι έγινε με την επικύρωση της συνθήκης. Όταν οι Ιρλανδοί ψήφισαν όχι είπαμε ναι συμφωνούμε με τη δημοκρατία αλλά μόνο όταν ψηφίζεται αυτά τα οποία εμείς υποστηρίζουμε. Αυτή είναι η δημοκρατία που υποστηρίζουμε. Ευχαριστώ. Καμάλ, damit wären die Stimmerklärungen zu Ευχαριστώ και κλείνει ε, ο κύκλος επεξηγήσεων ψήφου στο θέμα των εξωτερικών σχέσεων και ερχόμαστε στην έκθεση Μπροκ. Ο κύριος Άν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για μία ακόμα φορά θέλω να υπενθυμίσω τους συναντέλφους ότι το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και η Συνθήκη ο δεν είναι ακόμα σε ισχύ. Και κάθε άρθρο της έκθεσης Μπροκ ε, υπονοεί ότι αυτά τα, ε, είναι σε ισχύ, αλλά δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό είμαι κάπως καχύποπτο για το πώς προχωρούμε. Και βεβαίως ε, για την ε, ε, ψήφο που έγινε, για το δημοψήφισμα που έγινε στην ε, Ιρλανδία και το τελικό αποτέλεσμα. Διότι εδώ κάποιοι επιδιώκουν να ε, δημιουργήσουν ένα διπλωματικό σώμα. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει de facto αλλά δεν υπάρχει de jure. Από την άλλη ξέρουμε ότι όλοι έχουμε πρεσβευτές, οι χώρες μέλη έχουν πρεσβευτές στις διάφορες χώρες μέλη και τώρα θέλουμε να εισαγάγουμε μια νέα πρακτική και δεν, ε, δεν αντιδράει κανείς γιατί αυτή είναι η κοινή πρακτική εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι πραγματικά απίστευτος αν το σκεφτεί κανείς. Ευχαριστώ συνάδελφε Χέναν. Αυτή ήταν η μόνη επεξήγηση ψήφου στην έκθεση Μπροκ και τώρα προχωρούμε στην προετοιμασία της συνάντησης του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου. Δύο επεξηγήσεις ψήφου. Ο κύριος Μπολτσιτής. Ελπίζω να πρόφερα καλά το όνομά σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Υποστήριξα το ψήφισμα διότι θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για την επικείμενη συνάντηση σχετικά με το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο. Για τον λόγο λοιπόν αυτό, η ΕΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ηγηθούν ό,τι αφορά την εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχουν ανοιχθεί στο πλαίσιο των ε, G20. Δεν ε, χρειαζόμαστε μια στρατηγική σχέση μόνο με τις ΗΠΑ και αυτό ελπίζω να το λάβει υπόψη της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ τελευταία δήλωση του κ. Κάμαλ. Να ευχαριστήσω όλους σας για την υπομονή συμπεριλαμβανομένων και των διερμηνέων που έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Θα ήθελα να πω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Ε, έχουν ιδιαίτερη σημασία σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό στο διάλογο που εξάγεται όχι μόνο στο πλαίσιο της Διατρατικού Οικονομικού Συμβουλίου. Θα πρέπει να δούμε επίσης τι μορφή ηγεσία μπορούμε να προσφέρουμε. Και ένα από του καλύτερου τρόπου για να παροτρύνουμε τι οικονομίε μα, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο κρίση, είναι να διασφαλίσουμε πω ε, ε, προωθούμε το ελεύθερο εμπόριο. Με ανησυχεί το ζήτημα της κοινή ε, αγροτική πολιτική κάτι το οποίο πολλέ φορές ε, οδηγεί σε αύξηση του προστατευτισμού. Αν κοιτάξετε την κυβέρνηση Ομπάμα και του τελευταίου δασμού, που έχει υποβάλει στους Κινέζους νομίζω ότι οριστένουμε προς, τον προστατευτισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Καμάλ. Σας εύχομαι καλή όρεξη. Διακόπτουμε τις εργασίες μέχρι τις 15.00.